για τις αρμοδιότητες. Έχετε, Έχετε κάτι για το διαδικαστικό, κύριε Αγιάλα Σέντερ. Διαδικαστικό. Ακριβώς, πρόεδρε. Παρακαλώ, δώστε μας την δυνατότητα τώρα που μιλάμε με τους επιτρόπους. Έχουμε και κάποιο συγκρότημα με τύμπανο κρουσίες και που προέρχονται από τη λεγόμενη Βία Ντεμπουνιουέλ να μας ξυπνήσουν ίσως από το λίθαργο που ήταν. Ναι, καλά λέει ο Πρόεδρος. Όντως διαδικαστικό περνάμε λοιπόν στην ε, εγκριθήσα απόφαση σχετικά με, τα νέα, με τη νέα ατζέντα δεξιότητων για την Ευρώπη, δήλωση της Επιτροπής με την κυρία Μαριάννη Τάισεν. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, με μεγάλη μου ικανοποίηση εδώ στο Στασβούργο και σας παρουσιάζω το νέο θεματολόγιο για τις δεξιότητε που θα εθετηθεί και θα ανακοινωθεί επισήμω στον τύπο την Παρασκευή. Χαίρομαι που είμαι ήδη εδώ σήμερα μαζί σας για να συζητήσω μαζί σα τα βασικά στοιχεία του θεματολογίου αυτού. Οι δεξιότητε ε, είναι αντικείμενο μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλλει το θεματολόγιο στην υπόσχεση να δώσουμε αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τις θέση απασχόληση. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο. Συμβάλλατε ενεργά στη συζήτηση για τι δεξιότητε και τα προσόντα από τη φθεσινή έκθεση για να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνιστική αγορά εργασία για τον 21ο αιώνα τη κυρία Τζαβαλόβα μέχρι την έγκριση του ψηφίσματο φέτο για την πολιτική, ε, τις και την ε, πολιτική για τους νέους, Μάρικ Πλούρα και την έκθεση για και επαγγελματική κατάρτιση έκθεση Μαραγάλ και αυτά είναι απλώς μερικά στοιχεία, μερικές αυσοτοβουλίες σας. Έχουμε και κάτι άλλο. Χρησιμότατη ακρόαση της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Πολιτισμού που έλαβε χώρα τον Απρίλιο, όπου είχα συμμετάσχει μαζί με τον συνάδελφο Τίμπορ Ναυρασίτσου. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, οι δεξιότητες είναι ένα μονοπάτι προς την ευημερία. Οι σωστέ δεξιότητες δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αποκτήσουν ποιοτικέ θέσει εργασία και να εκπληρώσουν τελικά, να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό τους σαν ενεργοί πολίτες. ζει η οικονομία παγκόσμια και οι δεξιότητες καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τη δυνατότητα να προωθεί την καινοτομία. Η κατάσταση όμως στην Ευρώπη απαιτεί δράση. Ε, πάνω από 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν έχουν καλές ικανότητες ανάγνωσης, γραφής ή ψηφιακές δεξιότητες. Ένας στους τέσσερις ενήλικες δεν έχει περάσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν έχει πάρει προσόντα από δευτεροβάθμια. Πολλοί εργάζονται σε θέσεις που δεν ταιριάζουν με τα ταλέντα τους. Οι γυναίκες είναι το 60% των νέων αποφύτων, αλλά ο ρυθμός απασχόλησής τους είναι κάτω από αυτό των ανδρών. Ταυτόχρονα 40% των Ευρωπαίων εργοδοτών έχουν πρόβλημα να βρουν ανθρώπους με τις σωστές δεξιότητες. Και πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες για να δημιουργήσουν τη δική τους ε, επιχείρηση. Έτσι δε περαιτέρω, η ψηφιακή μεταμόρφωση αναδημορφώνει τον τρόπο ζωής μας, εργασίας μας και τον τρόπο επιχειρηματικότητάς μας και επίσης και τις ανάγκες που έχουμε σε δεξιότητες. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ελλείψεις σε ε, προσόντα υψηλά. Ε, ήδη το συζητήσατε αυτό με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Αβραμόπουλο, και παρά τα αποτελέσματα καλά για την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ε, είναι δεύτερη επιλογή για πολλούς. Με οι εθνικές και οι περιφερειακές αγορές εργασίας αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και δεν υπάρχει καλό ταιριάσμα αναγκών και εκπαίδευσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, το νέο θεματολόγιο για της δεξιότητας στην Ευρώπη εστιάζεται επί τριών τομέων προτεραιοτήτων. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα επίπεδα των δεξιοτήτων και να είναι οι δεξιότητες ανάλογες με τις ανάγκες αγοράς εργασίας. Άρα οι δεξιότητες και τα προσόντα θα είναι πιο εύληπτα και συγκρίσιμα διασυνοριακά μεταξύ διαφόρων οικονομικών τομέων θα είναι πιο προβλέψιμη η κατάσταση και θα υπάρχει καλύτερη κατανόηση των αναγκών σε δεξιότητε και προσόντα και τώρα και στο μέλλον. Χρειάζεται αύξηση των δράσεων. Δεν θέλουμε να μείνει κανεί πίσω. Γι' αυτό προτείνουμε μια βασική εγγύηση δεξιοτήτων. Είναι σύσταση προ τα κράτη-μέλη. Να συνεπιφέρουν του πόρου του, ούτω ώστε άνθρωποι με χαμηλά προσόντα να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τι αναγκαίε δεξιότητε που θα του βοηθήσουν να βρουν δουλειά. Να παραμείνουν στη δουλειά τους ή να βελτιώσουν την κατάστασή τους όσον αφορά την εργασία του Η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων θα διευκολύνει την κατασταση του οσον αφορα την εργασια του η αναθεωρηση του ευρωπαικου πλαισιου προσοντων θα διευκολυνει την κατασταση θα μπορούμε να συγκρίνουμε καλύτερα τις δεξιότητες και τα προσόντα. Έτσι, θα διευκολυνθεί κινητικότητα όσον αφορά τις μελέτες και την εργασία. Έχουμε ετοιμάσει και ένα σχέδιο για δεξιότητες που απαιτούνται σε διάφορους οικονομικούς τομείς. Θέλουμε να υπάρχει συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων, να εντοπίσουν τις ανάγκες σε δεξιότητες, να εντοπίσουν πρακτικές λύσεις. Αξιότιμα μέλη, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έρχονται στην Ευρώπη με πολλά προσόντα ποικιλία προσόντων μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομία μας. Για να διευκολύνουμε την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, προτείνουμε ένα εργαλείο για υπηκόστοι των χωρών να μπορούμε να εντοπίζουμε τις δεξιότητες που έχουν. Να τεκμηριώνουμε τα προσόντα τους. Να έχουμε μια εικόνα για αυτούς. Ποια είναι η επαγγελματική τους εμπειρία επίσης. Λοιπόν, ένα κοινό νήμα του θεματολογίου υπάρχει. Η ανάγκη να υπάρχει σύμπραξη παιδείας επιχειρήσεων όπως το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Νεολαία. Αυτές οι συμπράξεις, συνεργασίες, θα παίξουν κρίσιμο ρόλο, να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και να αλλάξει η νοοτροπία όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Άλλες δράσεις θα ακολουθήσουν την επόμενη διετία. Αργότερα φέτος θα προτείνουμε μια αναθεώρηση του πλαισίου Ευρώπας για την υποστήριξη της τεκμηριώσεως των προσόντων και δεξιοτήτων Χρειαζόμαστε ευφύ προσέγγιση για τις δεξιότητες και στηριζόμαστε στην υποστήριξή σας για να εγκριθεί γρήγορα αυτό όταν έρθει η ώρα. Ξεκινάμε και μια συμμαχία ψηφιακών δεξιοτήτων με εργασίες. Θέλουμε να μαζέψουν τα ταλέντα στον ψηφιακό τομέα. Όλοι, σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό θέλουμε. Για το 2017 έχουμε δρομολογήσει αναθεώρηση του πλαισίου ε, δεξιοτήτων του 2007 θέλουμε να ξεγχρονιστεί η επαγγελματική ε, κατάρτιση και προβλέπουμε πρωτοβουλία για την προσέλκυση των αποφύτων και να την παρακολουθούμε τους αποφύτους μάλλον, να δούμε πώς προχωράνε από την αποφύτηση στην αγορά εργασίας, ποια είναι η πορεία τους. Υπάρχουν πόροι ευρωπαϊκοί που μπορούν να βοηθήσουν να εφαρμόσουμε τις προτάσεις για την περίοδο 2014 μέχρι 2020 Έχουμε πάνω από 27 δισεκατομμύρια ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία για την στήριξη των δεξιοτήτων. Η ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται από το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε, το λαό μας. Η οικονομία του κόσμου αλλάζει γρήγορα και παίζει ρόλο η δεξιότητα του ανθρώπου. Έτσι θα είμαστε ανταγωνιστικοί και έτσι θα αναπτυχθούμε. Το θεματολόγιο των δεξιοτήτων δείχνει το πώς η Ευρώπη θα δώσει προστιθέμενη αξία στι δράσει των κρατών μέλων πώς θα κινητοποιηθούν οι διάφοροι φορείς. Μαζί, μαζί μπορούμε να ξεκλειδώσουμε το πλήρες δυναμικό της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, Επίτροπε. Και τώρα παίρνουμε στου ομιλητέ εκ μέρου των ομάδων. Ο κύριο Κάσα για δύο λεπτά. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, εμείς θεωρούμε θετική αυτή την πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο των Δεξιοτήτων. Έτσι θα γεφυρώσουμε κάποιες αποστάσεις, κάποιες διαφορές, οπότε και κάποιοι που το χρειάζονται θα μπορέσουν να προχωρήσουν όσον αφορά την ανάγνωση, τα μαθηματικά. Επίσης ε, νομίζω ότι είναι σωστό ότι δεν ε, ασχολούμαστε μόνο με τα ακαδημαϊκά, αλλά και τα επαγγελματικά. Πάρα πολύ καλά τα εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να θεωρηθούν προσόντα δεξιότητες ακριβώς όπως οι πανεπιστημιακοί τίτλοι και έτσι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές. Θα πρέπει να συνοηθούμε με επιχειρήσεις, με ιδρύματα, κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστήμια και έτσι να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε την ύλη και να είναι πιο κοντά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τα κράτη-μέλη να ενθαρρυνθούν να αξιοποιήσουν τους δάσκαλους και καθηγητές και αυτοί να αποκτήσουν τα προσόντα και δεξιότητες που χρειάζονται. Επίσης είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το καινούργιο θεματολόγιο γιατί διακρίνεται από ευελιξία και από προσαρμοστικότητα. Άρα έχει τις προϋποθέσεις να πετύχει ότι θέλουμε στην αγορά απασχόλησης που αλλάζει με ρυθμούς γρήγορους Άρα θα πρέπει να έχουμε στις πολιτικές μας ε, συνοχή, συνέπεια και στα κρατημέλη και για να πετύχουμε το στόχο μας να έχουμε ε, πρόσωπα τα οποία να μπορούν να διαβάσουν, να γράψουν, να μιλούν πάνω από μία γλώσσα, να μπορούν να είναι ε, συνηθισμένοι, εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά και έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην επιχειρηματικότητα. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Στάινρουκ, δύο λεπτά. Η εκπαίδευση είναι το μέλλον μας και πρέπει να το έχουμε το θέμα αυτό πρώτο στην ημερήσια μας διάταξη, το θεματολόγιο των καθηκόντων μας για τα χρόνια που έχουν περάσει, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις, ε, οι οποίες όμως είχαν μειωτική τάση και από αυτό ναι. βέβαια επλήγει το σχολικό σύστημα στην Ευρώπη και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ψηφιακής οικονομίας, ψηφιακές δεξιότητες στη, ε, στην Ευρώπη δεν είναι του ύψιστου επίπεδου. Ε, χρειάζεται λοιπόν μια επιτυχή στρατηγική, μια αποτελεσματική στρατηγική εκπαίδευση που συνεπάγεται τρία πράγματα. Πρώτον, δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση και με διδασκαλία των ψηφιακών δεξιοτήτων, γιατί όλοι χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις, να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να έχουν την αυτοπεποίθηση να τις υλοποιήσουν, να μπορούν δηλαδή να φτιάχνουν σχέδια για τη ζωή τους και με την πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία ως ε, όχι απλώς χρήστες αλλά ως παράγοντες. Δεύτερον, χρειάζεται η ανάπτυξη προφίλ ε, συνόλων δηλαδή δεξιοτήτων για τους νέους και σε σχέση με την κατάρτιση και την επαγγελματική απασχόληση ε, έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν οι δεξιότητες σε μια στρατηγική δεξιοτήτων. Χρειάζεται επίσης η διαβίου μάθηση η οποία θα παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις που είναι πολύ γρήγορες βέβαια και έτσι θα ενισχυθεί και η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται και μια στρατηγική αναγνώριση δεξιότητων και πιστοποίησή του. Πρέπει να θεσμοθετηθεί η διαβίου μάθηση. Φερρυπίν. Με μια εγγυημένη ελάχιστη απέτηση κάποιες αμοιβή γιατί δεν είναι δυνατόν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσφέρουν αυτή την πιστοποίηση χωρίς κάποια αμοιβή. Ευχαριστώ εκ μέρους τη ομάδα ΕΣΥΑΡΟ ο κύριος Κρασνοντέψκη. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Κυρία Επίτροπε, συμφωνώ με τους προαλήσαντες συναδέλφους ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση των δεξιοτήτων και άρα είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία σας. Επίσης, ας προσέξουμε το ότι δεν μπορούμε πλέον να ασχολούμεθα μόνο με το έλλειμμα που έχουμε στα επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την αύξηση της ζήτησης αυτών των ε, δεξιοτήτων, γιατί υπάρχει εδώ χάσμα μεταξύ των προσφερωμένων δεξιοτήτων και της ε, ζήτησης από πλευράς ε, αγοράς. Άρα θα πρέπει να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα και σύμφωνα με την σχετική έκθεση του 2015 έχουμε 25% ε, ε, των απασχολουμένων που είναι overqualified, έχουν ιδιαίτερα πολλά προσόντα και 27% που επίσης ε, έχουν τόσα πολλά προσόντα που δεν τα καλύπτει, δεν τους ικανοποιεί η δουλειά τους. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Η κυρία Ντλαμπάγεβα εκ μέρους των δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε επίτροπε, συνάδελφοι. Περιμένουμε ανυπόμονα την παρουσίαση του θεματολογίου για τις νέες δεξιότητες έτη δε περαιτέρω, διότι είναι βασικό θέμα που προσπαθούμε να προωθήσουμε με τους συναδέλφους μας της ομάδας των φιλελευθέρων. Αν μιλάμε για νέες δεξιότητες θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Είπατε ίδια κυρία Επίτροπε ότι πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχουν πρόβλημα να βρουν εργαζομένους με τα κατάλληλα προσόντα, κυρίως ε, ψηφιακά προσόντα. Θα πρέπει να έχουμε και όλα μεγαλύτερη κινητικότητα όσον αφορά το εργατικό δυναμικό. Η αναγνώριση των προσόντων και μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά τις γνώσεις στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι κάτι που απαιτείται. Προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού. Χρειάζονται αυτά. Είναι καθήκον μας να δείξουμε στους νέους ότι η αγορά εργασίας ε, λειτουργεί πραγματικά. Θα πρέπει να συνεργαστούμε ούτω ώστε η μαθητεία και η κατάρτιση, η τεχνική κατάρτιση για τους νέους να είναι κάτι πιο ελκυστικό. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην προετοιμασία μέσω της μαθητείας, μέσω της εργασίας, να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις προδιαγραφές της επαγγελματικής κατάρτισης και της παιδείας. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να γίνουν γνωστές οι ανάγκες ε, του αυριανού κόσμου. Αν η ευρωπαϊκή οικονομία θέλουμε να αναπτυχθεί περαιτέρω, τότε χρειάζονται όλα αυτά τα μέτρα. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την πρακτική σας προσέγγιση για το ανοιχτό σας πνεύμα στις συζητήσεις μας. Ελπίζουμε ότι αυτό το θεματολόγιο θα ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ο κύριος Πιμέντα Λόπες, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χρησιμοποιώντας σαν δικαιολογία τη μεγάλη ενεργία στην Ευρώπη, προσπαθούμε να πετύχουν το στόχο της Ευρώπης για το 2020. Δηλαδή βασικά υποθέτει ότι 25% του πληθυσμού του ευρωπαϊκού θα είναι άνεργο. Η διαβίου εκμάθηση είναι απλώς μια δικαιολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να κάνει την παιδεία και την κατάρτιση υπόδουλη όχι του λαού, αλλά υπόδουλη της ανάγκης των αναγκών ε, των επιχειρήσεων. Και έτσι αυξάνεται η κοινωνική διάκριση. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας πράγματι. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για να εισάγουμε ευελιξία μειώνοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων και εφαρμόζοντας νεοφιλελεύθερα προγράμματα. Δεν θέλουμε να γίνεται εκμετάλλευση των λαών, θέλουμε να δουλεύει ο κόσμο. Κυρία Τζιν πράσινη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και εγώ το εκτιμώ ότι έχουμε μπροστά μα τα έγγραφα. Ήταν καλό να είναι ενδελεχή η συζήτηση. Ξέρουμε όμω ότι έχουμε βασικές ελλείψεις όσον αφορά τι δεξιότητε. Το συζητήσαμε αυτό. Συζητήσαμε την πρόταση για την μπλε κάρτα και ξέρουμε ότι δεν είναι πρόβλημα μόνο του ψηφιακού τομέα αλλά και στη μηχανολογία. Ε, έχουμε τεράστια κενά εκεί στους μηχανικούς. Ελπίζουμε οι νέες προτάσεις να επανεξετάσουν το θέμα τα βασικά στοιχεία, βασικά προσόντα πρέπει να αναπτύσσονται κυρίως σε σχέση με το φύλλο ποια προσέγγιση ακολουθούμε. Σε μια πρώτερη έκθεση εξετάζαμε τις αλλαγές οικονομίες. Θέλαμε να είναι μια οικονομία πιο βιώσιμη με χαμηλότερη χρήση και εκπομπέ άνθρακος. Είχαμε διάφορες συστάσεις σε αυτή την έκθεση για τις δεξιότητες και ελπίζω να ληφθούν υπόψη αυτές οι συστάσεις τις προτάσεις που αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφορετικά, απλώς είμαστε καταδικασμένοι σε επανάληψη των εκθέσεών μας χωρίς να προχωρούμε. Ευχαριστώ. Τελευταία εκ μέρους των ομάδων. Η κυρία Ατζέ, η ευθύτη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Το 2011 προτείνατε το θεματολόγιο για τις ε, νέες δεξιότητες και αρμοδιότητες σε σχέση με την απασχόληση. Δεν έγινε τίποτα. Και κάναμε τις νέες μεταρρυθμίσεις σε Ιταλία, ε, Γαλλία, Ελλάδα και είδατε τι αποτέλεσμα πετύχαμε και ζητήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κινητικότητα των εργαζομένων. Αλλά σήμερα η μόνη κινητικότητα που υπάρχει στην απασχόληση είναι η εγκέφαλη, η εκροή των εγκεφάλων που οι άνθρωποι που φεύγουν δηλαδή, τη Βόρεια Ευρώπη. Άρα θα πρέπει κάτι να γίνει σε κινητικό επίπεδο γιατί ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων. Είπαμε ότι έγινε η αναθεώρηση αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί και τώρα το ξαναψάχνουμε. Άρα δεν υπάρχει επιλογή ε, επί της ε, ουσίας της πολιτικής. Κάτι που να είναι προς συμφέρον των εργαζομένων. Κάτι για αυτό που χρειάζεται η κοινωνία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό και τριάντα. Η κυρία Σάντερ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δεξιότητες. Οι δεξιότητες ε, συνιστούν σήμερα το στοιχείο κλειδί για να δώσουμε απάντηση στις βαθιτές μεταλλαγές που γνωρίζει η Ευρώπη και που χαρακτηρίζονται από πόλωση των συνθήκων ε, απασχόλησης με πολύ υψηλή δεξιότητα και δημιουργικότητα ε, θέση εργασία αφενό και πολύ χαμηλή κατάρτισης θέση εργασίας αφετέρου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε στο δυνατόν δεξιότητε δεξιότητες όλους τους Ευρωπαίους με ε, γνώση, τεχνογνωσία αλλά και ε, γνώσεις ζωής για να μπορούν να ενταχθούν στην επιχείρηση. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η κατάρτιση, η επαγγελματική κατάρτιση. Πρέπει να αναβαθμιστεί ανεξαρτήτως επίπεδου σπουδών και ανεξαρτήτως του σταδίου της ζωής στην οποία δίδεται αυτή η κατάρτιση στην, στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση στη διαβίου μάθηση. Εξασφαλίζουμε λοιπόν και μια πλατφόρμα αξιολόγηση των ε, δεξιοτήτων που θα είναι ένα κατάλληλο βήμα ασφαλώς, πρώτο βήμα όμως που ταυτόχρονα θα πρέπει να δίνει περισσότερα ενάψματα για απασχόληση κυρίως για τους πιο ευάλωτους, εκείνους που δεν έχουν τις δεξιότητες ώστε να ε, διεκπαιρεώσουν τις ε, αιτήσει τους μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας. Θα ήθελα λοιπόν και να χαιρετήσω την πρωτοβουλία σας κυρία Επιτροπή αλλά και να επιμείνω ότι χρειάζεται και τα κράτη-μέλη να στρατευτούν προς την διακατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαντέρ. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Σάνι. Κύριε Σάνι, έχετε το λόγο 30 δεύτερα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, Έχουμε, έχω να ρωτήσω λοιπόν το εξής για τη στρατηγική 2020. Όσο τμήμα της στρατηγικής αυτής έχουμε ορίσει μια ατζέντα και για τις δεξιότητες Ωστόσο έχει ξεκινήσει κάποια βήματα η κυβέρνηση Ορμπάν η οποία αντίκειται σε αυτά τα οποία ορίζει το θεματολόγιο. Η κυρία Σάντερ για να απαντήσει 30 δεύτερα. Αγαπητέ συνάδελφε, πιστεύω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη την ανάγκη να επεξεργαζόμαστε νέα, νέες λύσεις για τις δεξιότητες και την κατάρτιση στη χώρα μου, τη Γαλλία. Η κυβέρνηση όρισε ως προτεραιότητα την κατάρτιση τουλάχιστον στα λόγια. Ταυτόχρονα όμως έλαβε μέτρα τα οποία αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και ιδίως τους, ε, τα χειρονακτικά επαγγέλματα από το να ελκύσουν ε, μαθητευόμενους. Νομίζω ότι πολλά βήματα πρέπει να γίνουν στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα στη δική μου τη χώρα, τη Γαλλία. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Σίλβια Κώστα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκτιμώ πολύ που ήδη η Επίτροπος η κυρία Τάισεν παρουσίασε τον θεματολόγιο για τις δεξιότητες στην Ευρώπη κυρία Τάισεν για να, αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα με τη χρήση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ελπίζω και το αίτημα που είχα προωθήσει σαν εκπρόσωπο τη Επιτροπή Πολιτισμού στη κοινή συνεδρίαση με την απασχόληση να επεξεργαστούμε το στόχο συνεννόηση με τον Επίτροπο κ. Ναύρασιτ για ολοκληρωμένη ολιστική προσέγγιση στα πλαίσια τη διαβίου εκμάθηση. Υπάρχει δεν υπάρχει τέριασμα μεταξύ των δεξιοτήτων προσφέρονται και εκείνων που ζητούνται. Πρέπει να ενισχύσουμε τι ψηφιακέ δεξιότητε, αλλά και τι βασικέ αρμοδιότητε των πολιτών και την υψηλή εκπαίδευση. Να προωθήσουμε τη συμμαχία τη γνώση και τη συμπράξεω μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων με τι επιχειρήσει, με την έρευνα, για να προωθήσουμε τον τομέα τη παιδεία, εργασία και καινοτομία, αυτή την αλυσίδα. Και επίση ε, μαθητεία και επαγγελματική κατάρτιση. Χρειάζεται να είναι ποιοτική η εκπαίδευση εκπαίδευση, η να υπάρχει συγκρισιμότητα των δεξιοτήτων και θέλουμε να γίνονται σωστές επιλογές από τους ανθρώπους για την καριέρα τους. Χρειάζεται κάποια βάθυνση η πρόταση για το Skills Guarantee για να δώσουμε προσωπικές δεξιότητες στους ανθρώπους, όπως και αναθεώρηση του πλαισίου, που, δηλαδή να συμπεριλαμβάνουμε καλύτερα τι άτυπε και μη επίσημε δεξιότητε. Βλέπω με χαρά ότι στι προγραμματισμένε δράσει του θεματολογίου τον Ιούνιο ξεκινά ένα εργαλείο αναγνωρίσεω των δεξιοτήτων εκείνων που έρχονται από τρίτε χώρε Είναι ένα μέτρο το οποίο είχαμε ζητήσει και για να προωθήσουμε και του διαδρόμου τη παιδεία για πρόσφυγε φοιτητέ στα πανεπιστήμια και στα ευρωπαϊκά σχολεία. Θα ήθελα να καταλάβω πώ το βλέπετε εσεί. Πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα στη συγκρισιμότητά τους και την κινητικότητα και των φοιτητών των πανεπιστημίων και εκείνων που είναι στην επαγγελματική κατάρτιση. Κλείνοντας, πιστεύω ότι είναι επίσης σημαντικό να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα της ενισχύσεως διαφόρων μέσων κατάρτισης των διδασκάλων και των κατατιστών εκείνων που κάνουν την κατάρτιση ε, μέσω πλατφορμών όπως είναι το e-teaching, ηλεκτρονικά δηλαδή. είναι η κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συμφωνούμε πάντοτε πως υπάρχει ανάγκη να αναβαθμιστούν και να προσαρμοστούν ε, οι δεξιότητες των εργαζομένων με βάση και τις εξελίξεις τεχνολογίας και τις ε, ανάγκες της αγοράς, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να υπαχθούν στα ιδιωτικά συμφέροντα αυτές. Ε, δεν μπορεί να ανεχθούμε ευελιξία και έκθεση σε τέτοιους κινδύνους των εργαζομένων. Θα πρέπει η επαγγελματική κατάρτιση και η μαθητεία να προσφέρουν ταυτόχρονα και κατάλληλη αμοιβή, όχι εκμετάλλευση. Δεν είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας να εκτεθούν στην εκμετάλλευση των επιχειρήσεων οι εργαζόμενοι. Ο καλύτερος τρόπος είναι να τους προσφερθεί η κατάρτιση και η μαθήση ε, με ολιστικό τρόπο. Και είναι βέβαια διαβίου διαδικασία που εμπλουτίζει τον άνθρωπο για να ωφεληθεί ολόκληρη η κοινωνία από αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αρέντ, και ένα λεπτό. Επίτροπε, συνάδελφοι, δεξιότητες. Αυτή είναι η νέα μαγική λέξη που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Όλοι, όλοι λατρεύουν ε, αυτή τη ε, λέξη, του τις νέες δεξιότητε, να, να βάλουμε μια φύσα με χαμογελού ανθρώπου και, και όλοι μαζί να φωνάζουν νέες δεξιότητες. Μα τι πάνε από αυτό και πώ ακούγεται ε, από τους νέους, από τους νέους που δεν έχουν δουλειά, τι θα τους δώσει, θα τους δώσει κάποιες ευκαιρίες. Μπάς και είναι μια στρατηγική, να τους δημονοποιήσουμε επειδή είναι άνεργοι. Συμπαθάτε με, μπορεί να έχετε τρία πανεπιστημιακά πτυχία, ένα μεταπτυχικό τίτλο, αλλά να μην έχετε ε, τις κατάλληλες δεξιότητες για να βρείτε δουλειά. Εάν θέλετε αυτό το θεματολόγιο να πετύχει ουσιαστικά, θα πρέπει να κάνετε κάτι για τα εκπαιδευτικά συστήματα, να λάβετε υπόψη τις επιθυμίες τις ανάγκες των φοιτητών και μαθητών και ένα πρόγραμμα επενδύσεων το οποίο να δημιουργεί τις θέσεις απασχόλησης όπου θα κολλάνε αυτές οι νέες δεξιότητες οι οποίες θα πρέπει από ένα σύνθημα να είναι κάτι το αυτό που να κάνει κάτι για τους Ευρωπαίους στην καθημερινή του ζωή αλλιώς δεν πετύχαμε στη δουλειά μας και στο έργο μας. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας από τον κύριο Σούλτσε. Τη δέχεστε. 30 δεύτερα κύριε Σούλτσε. Κύριε Ρέντκε, εγώ έχω μόνο ένα πτυχίο μηχανικός. Δεν δυσκολεύτηκα όμως να βρω μετά τις σπουδέ μου ε, μια θέση εργασία. Εσείς λέτε ότι άνθρωποι με τρία πτυχία και ένα μάστερ δεν καταφέρουν να βρουν δουλειά. Δεν καταλαβαίνω το επιχείρημά σας. Νομίζετε δηλαδή ότι δεν χρειαζόμαστε τις ε, νέες δεξιότητες, αυτή είναι η απόψη των πρασινών. Mm. Κυρία Ρέντκε, στα γερμανικά. Ναι, πηγαίνετε λίγο στην Ισπανία να, δει, να δείτε υπάρχουν άνθρωποι με τρία πτυχία και καμία δουλειά. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό, στο ότι δεν χρειαζόμαστε ε, θεματολόγιο νέων δεξιοτήτων, αλλά ένα πρόγραμμα που θα δημιουργεί θέσει εργασία για αυτού του νέου που έχουν την κατάρτιση. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Βεβαίω και χρειαζόμαστε τι δεξιότητε, αλλά ταυτόχρονα και άλλε δραστηριότητε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να δώσουμε προοπτικέ σε αυτού του νέου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι νόημα έχει να κουβεντιάζουμε γι' αυτό το θεματολόγιο των δεξιοτήτων. Ο πρόεδρος της Τουρκίας που είναι υποψήφια χώρα για ένταξη λέει ότι οι γυναίκες που δεν κάνουν παιδιά είναι ε, μισοί άνθρωποι. Όμως τι είναι αυτό να έχει κανείς ε, δουλειά και παιδιά για να έρχεται τα δύο μα δεν σέβονται τις γυναίκες σε εκείνη τη χώρα το μόνο που του ενδιαφέρει είναι η αναπαραγωγική δυνατότητα και το να φροντίζουν και να καθαρίζουν το σπίτι και τον άντρα τους. Οπότε θα πρέπει να δούμε το πόσο είναι τεράστια η συμβολή των ε, γυναικών στον πολιτισμό, τις σουφραζέντες, την Μαρία Κιουρί, ε, τους ε, λογοτέχνες, τι έγινε στους δύο πολέμους, τι γίνεται τώρα, γιατί περιθούν γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις. Τι γίνεται, υπάρχουν κάποιοι φεμινιστές και φεμινίστριες που υποστηρίζουν εκείνη τη χώρα. Ελπίζω οι Αγγλίδες αυτό να το συνειδητοποιήσουν. Σας ευχαριστώ και σας ε, υπενθυμίζω ότι βεβαίως έχετε το ελεύθερο να μιλάτε για το θέμα που σας ε, απασχολεί, αλλά ξέρετε ότι δεν ήταν το θέμα μας ε, στο θεματολόγιο των δεξιοτήτων η συζήτηση για την Τουρκία. Αλλά εσείς αποφασίσατε τι θέμα θέλετε να προβάλλετε. Η κυρία Σόιτροβα, ένα λεπτό και 30 δεύτερα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για την παρουσίαση που έκανε για την ώρα δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία συγκεκριμένα όσον αφορά το θεμετολόγιο. Αυτό που θα ήθελα να πω εδώ είναι να θέσω κάποια σημεία, κάποιες ερωτήσεις, να θέσω κάποιες προσδοκίες που έχω να παρουσιάσω όσον αφορά το ευρωπαϊκό θεματολόγιο των δεξιοτήτων. Αυτό το θεματολόγιο είναι απαραίτητο. Αναφερθήκατε και ποια ήταν η αφετηρία του θεματολογίου. Δεν θέλουμε μειώσουμε τον αριθμό των μαθητών. Ε, μάλλον θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο. 20% των νέων δεν φτάνουν στο να ολοκληρώσουν ε, την βασική τους εκπαίδευση. Λοιπόν, όσον αφορά την αφετηρία του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων, αυτή η αφετηρία εδράζεται επί νέων ερευνών. Θα χρησιμοποιήσετε τις έρευνες ε, του EPS που έχουμε, θα έχουμε ή ξεκινάτε αποκλειστικά από αποτελέσματα δικών σας προτέρων εργασιών. Φαντάζομαι ότι το θεματολόγιο των δεξιοτήτων θα έχει σαν στόχο τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων. Υποθέτω επίσης ότι θεματολόγιο επίσης θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δεν είναι δυνατόν να περιοριζόμαστε μόνο στις ανάγκες της αγοράς, λησμονώντας την ανάγκη να εξασφαλίσουμε τις βασικές γνώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζουμε αυτές τις ε, προτάσεις για το θεματολόγιο των δεξιοτήτων ε, όλα αυτά τα οποία αφορούν το skills guarantee και όσον αφορά την αξιολόγηση του πλαισίου των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Θα πρέπει να βελτιωθεί όμως η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει οι πιο ευάλωτοι να είναι εύκολο να έχουν πρόσβαση. Να δούμε τις προτεραιότητες, τι με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων, αξιολόγηση των επαγγελματικών συστημάτων, ε, ε, όσον αφορά επίσης και τις δεξιότητες και προσόντα μεταναστών και προσφύγων τα σήμερα συζητούμενα μέτρα να είναι συμπληρωματικά στις προσπάθειες για επένδυση και επενδύσεις τέλο πάντων και όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα γιατί χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αυτή η υπόθεση των νέων δεξιοτήτων δεν θα αρκέσει. Ε, ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Κούνεβα παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανεξασφάλιση εργασία για το 75% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού μέχρι το 2020 είναι κεντρικό στόχο τη Ευρώπη 2020, τότε οι ήδη αποτυχημένε πολιτικέ και τα προγράμματα κατάρτιση δεν λύνουν το πρόβλημα τη ανεργία. Ναι, να αναβαθμιστούν οι δεξιότητε, αλλά με ποιο στόχο σίγουρα όχι την αποκλειστική εξυπηρέτηση των συμφερόντων της αγοράς αλλά να έχουν όλοι οι πολίτε καλύτερα εφόδια για τη ζωή μέσα από ισότιμη πρόσβαση σε δημόσια εκπαίδευση υψηλή ποιότητα Η τυφλή προσαρμογή της εκπαίδευσης στην αγορά εργασία η εμπορευματοποίηση της και η αποβάθμιση των κλασικών σπουδών δεν έχει καμία σχέση με το ρόλο της που αποσκοπεί να χτίσει ελεύθερε προσωπικότητε. Γι' αυτό η ατζέντα των νέων δεξιοτήτων να αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων σε γνώσει και προσόντα και όχι μόνο στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ιζαμπέλα Αντινόλφη έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχει αυτή η αιμονή με τις δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτυχθούν και αυτό θεωρείται ότι ε, κάνει τους ε, ανθρώπους σαν μια πηγή, ε, σαν ένα κεφάλαιο που κανείς πρέπει να καταλευθεί και αυτή είναι μια προσέγγιση λανθασμένη. Θα πρέπει επομένω να δούμε το ότι απέτυχε στην Ιταλία και στην ε, Γαλλία όπως αποδείται από τις μεταρρυθμίσεις αγοράς εργασίας. Ε, είναι πάρα πολύ ευάλωτοι τώρα οι νέοι και γίνονται αντικείμενα οι νέοι που θα πρέπει να τα περιβάλλουμε με κάποιες τέτοιε τέτοιες ε, δεξιότητες γιατί έτσι δεν γίνεται τίποτα για οικονομική ανάπτυξη. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, το εργαλείο που είναι η εγγύηση για τους νέους και θα πρέπει να δυσυντούσουμε ότι δεν έχουμε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει ανεργία για τους νέους, ιδίως στον ε, Νότο. Θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να εγκατέλειψουμε αυτά τα προγράμματα που επιβάλλονται από τα πάνω και να ληφθούν υπόψη ιδιωτικίες και πραγματικές ε, ανάγκες των πολιτών. Κύριε Φαντερ Κέντελάρ για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι ανάγκη νομίζω να σας υπενθυμίσω το, τη στρατιά αυτή των νέων Ευρωπαίων που είναι άνεργοι στις κάτω χώρες. Μπορεί τα στοιχεία σε σχέση με κάποιες νότιες χώρες ε, της Ευρώπης ε, και ιδιαίτερα της Μεσογείου να είναι ισχνά. Αλλά έχουμε πάλι μεγάλο πρόβλημα με νέους, ιδιαίτερα από οικογένειες μεταναστών ή εν πάση περιπτώσει που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας με υψηλή όμως κατάρτιση και παραμένουν χωρίς τις εργασίες. Γι' αυτό χρειάζεται αυτό το θεματολόγιο κυρίες και κύριοι γιατί δίνει απαντήσεις στα προβλήματα που εντόπισα μόλις τώρα. Έχουν κατάρτιση, έχουν δεξιότητες, έχουν ταλέντα οι άνθρωποι αυτοί και πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για τους ίδιους αλλά και για τον κάθε πιθανό εργοδότη να προσδιοριστεί αυτό το ε, αυτή η βαλίτσα που θα έχουν μαζί τους αυτό το ε, μπαγκάζι που θα τους συνοδεύει για να ξέρουν πώς μπορούν να το αξιοποιήσουν. Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι δεξιότητες ανοίγουν νέε πρωτοβουλίες για να μην χάνονται οι νέοι, να μην τους λησμονεί το σύστημα. Το Europass είναι ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί με θέσεις εργασίας στις ε, ανάγκες και τις ικανότητες του καθενός. Μια στρατηγική λοιπόν νέα για τις δεξιότητες που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των νέων συνθήκων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ουλσκό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε για αυτό το νέο θεματολόγιο των δεξιοτήτων είναι ένα κομμάτι της δουλειάς που ξεκινήσατε παλιά. Θέλετε να εξασφαλίσετε ότι τα προσόντα είναι πιο συγκρίσιμα μεταξύ κρατών μελών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τους νέους μέσω, του, μέσω της εγγύσεως για τους νέους. Εκείνους που ψάχνουν για δουλειά στην αγορά εργασίας, εκείνους που χρειάζονται περισσότερο την υποστήριξή μας. Αλλά ανησυχώ για κάτι. Ανησυχώ για την άποψη που αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα. Είναι κάτι που διαπνέει την ανακοίνωση. Εξαρτάται από τους επιχειρηματίες να ανταποκριθούν στην αλλαγή της κοινωνίας, να αντιμετωπίσουν θέματα ανασφάλειας περίπλοκων συνθήκων. Η επιχειρηματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά αν είναι να λύσει τα πάντα που περιγράφονται επιχειρηματικότητα δεν είναι υπερβολικό, δεν πάει πολύ μακριά. Νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι η επιχειρηματικότητα να είναι εφημισμός για την αυτοαπασχόληση ουσιαστικά που παρουσιάζεται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χούντης, παρακαλώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η νέα ατζέντα δεξιοτήτων που μας παρουσιάσατε μέσα στο νεοφιλελεύθερο κυρίαρχο εργασιακό πλαίσιο δεν διασφαλίζει πλήρη εργασιακά δικαιώματα αλλά απορριθμίζει περαιτέρω τι εργασιακέ σχέσει οδηγεί στη μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση εμπλέκει τι επιχειρήσει όλο και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία και εν τέλει ισχυρίζεται ότι για το φαινόμενο τη μετανάστευση των επιστημόνων από την ελλάδα και την ευρώπη φταίει το γεγονό ότι δεν υπάρχει καταρτισμένο επιστημονικά και εκπαιδευμένο προσωπικό. αυτή η δέσμη μέτρων κυρία επίτροπε είναι καταδικασμένη όπω και η συνολική σα πολιτική. δεν ενδιαφέρεστε για τον εργαζόμενο ενδιαφέρεστε για τα κέρδη των επιχειρήσεων. οι γάλλοι λοιπόν εργαζόμενοι και η νεολαία που έχουν βγει στους δρόμους τα βελγικά συνδικάτα που απεργούν το 25% των ανέργων στην ελλάδα το 40% των νέων ανέργων στην ελλάδα δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα από αυτές τις προτάσεις. αγωνίζονται για να ανατρέψουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε το λόγο έχει ο συνάδελφο Σούλτσε για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συμφωνώ με την πρόταση για το θεματολόγιο δεξιοτήτων γιατί μπορεί να δώσει απαντήσεις σε σχέση με την αγορά εργασίας και το συνδυασμό των δεξιοτήτων. Σε όλη την Ευρώπη μπορούμε να έχουμε αναγνώριση δεξιοτήτων και μια ενιαία αντίληψη για αυτές. Και έτσι μπορούμε να ανοίξουμε μια αγορά σε όλη την Ευρώπη, χωρίς σύνορα. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει καλή, μεγαλύτερη κινητικότητα σε σχέση με τους πτυχιούχους και ανάλογα με την κατάρτιση. Η μαθητή επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το διαδικό σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να την ενισχύσουμε αυτό πιστεύω ότι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω πρέπει να εμπνευστούμε από μοντέλα βέλτιστων πρακτικών, ώστε να δεχθούμε ο ένα από τι επιτυχίε του άλλου. Η επιτυχη εκπαίδευση όμω, η καλύτερη εκπαίδευση όμω, δεν οδηγεί απαραίτητα σε μια ασφαλή θέση εργασία. Το πρωτοαρχικό καθήκον για την βασική πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανήκει στο κράτο. Πρέπει να την προσφέρει λοιπόν το κράτο αυτό και να μην εγκαταλείπει τους πολίτες του ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Μετά και με μια στέρεα βάση από τη βασική εκπαίδευση μπορεί ο πολίτης να προχωρήσει στην περαιτέρω κατάρτιση. Η πρόταση σας κυρία Επίτροπε έχει την πλήρη υποστήριξή μου. Ευχαριστώ. Γκουτιέρες. Πρόεδρε, ε, κυρία Επίτροπε, θα υποστηρίξουμε αυτούς του στόχου συμφωνούμε, αλλά όχι για τα μέσα που διαλέξατε γιατί θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Υποστηρίζουμε το στόχο που θέσατε, γιατί κάτι θα πρέπει να στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα που έχουμε φτάσει σε ρεκόρ ενεργεία των νέων και λένε τις άντρες κατά των επιχειρηματών ότι δεν βρίσκουν τον κόσμο που χρειάζονται με σωστές ε, δεξιότητες και 50% των ε, μακροχρόνων ανέργων δεν έχουν την κατάρτιση που θα ενσύγουν τη στατιστική. Όμως δεν ωφελεί απλά έτσι ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο να υλοποιηθεί από τα κράτη-μέλη όπως τους ε, έρχεται. Χρειαζόμαστε αυθεντική εγγύηση και ε, πραγματική χρηματοδότηση, όχι απλώ συντονισμό. Χρειάζεται καλύτερη κατάρτιση για να σταματήσουν να υπάρχουν όλα αυτά τα κενά, τα χάσματα ε, για τα ψηφιακά, για μεταξύ των γενεών θα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε όλους και τους νέους και τους συνταξιούχους και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την απασχόληση και να υπάρξει αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των πόρων του να πάει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλιώ δεν θα υπάρξει πρόοδος. Ενάμεση λεπτό. Κυρία Κλούν. Ναι, ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες των όσων ανακοινώσατε, όπως είπε και ο προελής σας. Και εγώ θα πω ότι οι 20% των νέων είναι άνεργοι, 40% των εργοδοτών δεν βρίσκουν αυτούς που θέλουν τις καταρτήσεις που θέλουν και πάρα πολλοί από τους μεγάλους ανέργους δεν έχουν τις καταρτήσεις που χρειάζεται και όλα αυτά τα λέγαμε για τα μέσα της 1990 ότι το 50% των νέων δεν είχαν ε, δουλειά και δεν είχαν τις κατάλληλες δεξιότητες άρα μία από τα ίδια άρα θα πρέπει κάτι να κάνουμε με αυτό το θεματολόγιο να δούμε τι θα γίνει με εκπαίδευση, με κατάρτιση τόσο σημαντικά άρα θα πρέπει να εμπλακεί εδώ ε, και ο κλάδος της ε, βιομηχανίας αλλά και των εργοδοτών δεν αρκεί να γκρινιάζουν και να γονομοδοτούν πρέπει άμεσα να εμπλακούν και να υπάρξει επομένω σωστή χρηματοδότηση και από αυτού γιατί είναι προ το συμφέρον τους να εξελιχθούν και να αποκτήσουν δεξιότητε οι εργαζόμενοι. Μπράβο για όσα είπατε και μπράβο για τα 27 δις που θα δώσει το κοινωνικό ταμείο. Και ελπίζουμε ότι όλα τα κρατημέλη να συνεργαστούν να εκμεταλλευτούν αυτή την πρικοδότηση και να έχουν τα κατάλληλα προγράμματα για τις κατάλληλες δεξιότητες, αλλά βέβαια χρειάζεται ποιότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιδί, γιατί είπαμε οι 70 εκατομμύρια Ευρωπαίων που δεν ξέρουν όπως χρειάζεται αριθμητική ανάγνωση, γραφή. Άρα φυσικά πρέπει να και για την πρωτοβάθμια παιδεία. Και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται το νέο είδος οικονομίας για τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει και μεταξύ των εργαζομένων. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτής της νέας στρατηγικής. Αυτή την εποχή <coughs> δεν αρκεί να έχει κανείς αποκτήσει δεξιότητες μία φορά στη ζωή του ε, δεδομένου ότι οι συνθήκες, η τεχνολογία αλλάζουν τόσο γρήγορα πρέπει κανείς να θέσει να προσαρμόζει την μαθητεία του και να αποκτά νέες δεξιότητες διαρκώς. Και αντίστοιχα βλέπουμε ότι πολύ συχνά και ο εργοδότης δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό στη διάθεσή του. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε περισσότερο στα σχολεία και ιδιαίτερα να ενθαρρύνουμε του εργοδότε ώστε να προσφέρουν θέσει εργασία Τα σχολεία θα πρέπει να συνεργάζονται και με τα επαγγελματικά Ινστιτούτα ώστε να καταρτίζεται ένα προσωπικό ε, που ζητάει η αγορά. Επίσης η εκροή εγκεφάλων ή καλύτερα εργατικού δυναμικού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μέσα που, ώστε να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η νέα αυτή πρόταση, το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες είναι ευπρόσδεκτο και σας συγχαίρω κύριε Επίτροπε. Είναι όντως απαραίτητο για τον Ευρωπαίο πολίτη ο οποίος μπορεί χάρη στο εργαλείο αυτό που παρουσιάζεται να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος αλλάζει διαρκώς, πρέπει να μεριμνήσουμε για τους νέους, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και τις ανάγκες των εργοζομένων οι οποίοι θα χρειαστεί να προσαρμόσουν την, ε, τις δεξιότητές τους σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους. Καλό θα είναι να μην αναγκάζεται κανείς να παραμένει σε μια θέση εργασίας η οποία δεν αντιστοιχεί στο ταλέντο, στη φιλοδοξία του, στις δεξιότητές του. Πρέπει να εξασφαλίσουμε συνθήκες απασχόλησης που θα καλύπτουν τις ανάγκες των νέων από 20 ετών μέχρι και 64, 65 ετών. Πρέπει να υποστηρίξουμε τη μάθηση, τις ψηφιακής δεξιότητες και να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν και να δημιουργηθούν νέες εργασίες. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση, στη διαβίου μάθηση. Για όλους τους νέους. Θα συστήσουμε φαντάζομαι τις λεπτομέρειες αργότερα και θα μπορέσουμε να βρούμε και νέε δυνατότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό για την κυρία Λιμπάσικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την Επίτροπο Αναφερόμασταν στις δεξιότητες. Πρέπει να διερωτηθούμε όμως πρώτα ποια είναι η θέση της παιδείας στην κοινωνική ζωή. Η ποιότητα της παιδείας πρέπει να προσμετράται όχι από την ετοιμότητα κανείς να περάσει διαγωνίσματα, αλλά πόσο καλά είναι προετοιμασμένος κανείς για τη ζωή του. Υπάρχουν άλλες δεξιότητες που απαιτούνται, οριζοντίου φύσεως, αλλά και κοινωνικά και πνευματικά προσόντα χρειάζονται. Και Πρόεδρε πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρηματίες και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στην ίδια την παιδεία θα πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί, θα πρέπει επίσης να αναλάβουν την υποχρέωση επιχειρηματίες να δημιουργούν και θέσεις για τους νέους. Μετά θα πρέπει να αλλάξουμε μεθόδους και προγράμματα μαθημάτων και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το άτυπο μονοπάτι προς την εκπαίδευση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως είναι το πρόγραμμα Erasmus+, ούτως ώστε να εντατικοποιήσουμε την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και για τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί σε κάποια κράτη-μέλη και εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσης να λαμβάνονται υπόψη. Λοιπόν, να σέβεστε το χρόνο, έχουμε πάρα πολλά θέματα και ο χρόνος δεν είναι ε, άπειρος. Συνάδελφε Μούρεζαν, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σε 20-30 χρόνια οι περισσότερες θέσεις θα είναι σε κατηγορίες και θα πετούν προσόντα που δεν δεν υπάρχουν σήμερα. Όπως σήμερα εν συγκρίση με το τι γινόταν πριν 20-30 χρόνια. Και θα έχουμε ακόμα ταχύτερες τεχνολογικές αλλαγές στις επόμενες δεκαετίες. Ο τρόπος που θα εργάζεται ο κόσμος, θα προσλαμβάνεται ο κόσμος και πώς θα επιχειρεί θα είναι εντελώς διαφορετικό στο μέλλον από ό,τι σήμερα. Και η ταχύτητα θα αυξάνεται. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να εξοπλίσουμε τους νέους της Ευρώπης με σωστές δεξιότητες για να έχουν πρόσβαση στις μελλοντικέ θέσεις απασχόλησης. Συζητούμε το διαδίκτυο, την ψηφιακή ενιαγορά. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι κάτι που γίνεται προσωπικό. Εκεί αισθάνεται ο κόσμο ότι κάνει κάτι η Ευρώπη για αυτού, στον ψηφιακό κόσμο. Θα πρέπει οι οργανώσει των νέων να συμμετέχουν περισσότερο στη σύνταξη νέων προτάσεων για την απασχόληση. Η ψηφιακή ε, παιδεία θα πρέπει να είναι βασική δεξιότητα που θα αποκτάτε από πολύ νωρί και θα τελειοποιείται κατά τη διάρκεια τη ζωή. Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε εθνικό επίπεδο πρέπει να προσαρμοστούν δεόντω. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το εκπαιδευτικό του σύστημα ανταποκρίνεται στι ανάγκε τη αγορά. Δεν θα πρέπει να μείνουμε πίσω στην ανταγωνιστικότητα στον κόσμο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση ότι θα ανταποκρίνεται ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώση στι ανάγκε των νέων. Πρέπει να έχουμε κατάλληλο πλαίσιο, να παρέχουμε κάθε είδους βοήθεια στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να εξυγχρονίσουμε τα συστήματα παιδείας. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό επόμενος, παρακαλώ. Η επόμενη μάλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση διαβίου δεξιότητες. δεξιότητε δεξιότητες όσον αφορά το χώρο εργασίας και τη ζωή. Πρέπει να ετοιμάσουμε μια γενιά νέων που θα έχει κίνητρο. Θα έχει δεξιότητες, δημιουργική σκέψη, επιχειρηματικότητα, δυνατότητα να ηγούνται και να δημιουργούν δυνατότητες, δυναμικό, να είναι τολμηροί όσον αφορά τις λύσεις των προβλημάτων και να είναι και υπεύθυνοι πολίτες. Καλή λοιπόν η πρόταση. Θέλουμε οι νέοι να προετοιμαστούν να ζήσουν σε έναν κόσμο που αλλάζει τάχιστα, που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε σήμερα. Τι ξέρουμε όμως ότι ο μελλοντικός κόσμος θα είναι όλο και πιο ε, ψηφιοποιημένος και συνδεδεμένος με το διαδίκτυο. Λοιπόν, η ψηφιακή εκπαίδευση είναι βασική προϋπόθεση. Πρέπει ε, να εξοπλίσουμε τους νέους όμως να έχουν κριτική σκέψη και ψηφιακή περιέργεια που είναι απαραίτητα αυτά. Να μην γίνουν μόνο χρήστες τεχνολογίας, αλλά ενεργοί πολίτες σε μια συνδεδεμένη κοινωνία μέσω διαδικτύου. Η ραχοκοκαλιά του θεματολογίου των δεξιοτήτων πρέπει να είναι η παιδεία για το συνέστημα του πολίτου. Χρειάζεται ε, επίσης και μια εκπαίδευση για κάθε μορφή γνώσης με στο δικτύο. Ευχαριστώ η κυρία Πάουνοβα για 1,5 λεπτό. Κυρία Επίτροπε, οι απαραίτητε δεξιότητες για να πετύχει κανείς ε, είναι στα πλαίσια μιας ένωσης προοδευτικής και ανταγωνιστικής, οπότε είναι πολύ θετική η πρόταση σε 40% του πληθυσμού έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, όμως μόνο ένας εις τους τέσσερις εργοδότες καταφέρνει να βρει τις δεξιότητε που θέλει σαν εργαζόμενο που χρειάζεται, άρα πιστεύω ότι χρειάζεται μια άλλη ε, ομοιογενής προσέγγιση και πιο αποφασιστική πολιτική ηγεσία θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε ηλεκτρονικές ε, ε, δεξιότητες γιατί 90% των εργασιών στο μέλλον θα χρειάζονται γνώσεις πληροφορικής όμως ε, τώρα μόνο το 1 τρίτο των Ευρωπαίων έχουν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο χωρίς να λάβουμε υπόψη για το ότι δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς τι μορφή θα έχουν οι δουλειές στο μέλλον άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε το θέμα της αναγνώρισης των ε, ψηφιακών δεξιοτήτων ε, γιατί οι δεξιότητες δεν πρέπει μόνο να βοηθούνται αλλά θα πρέπει να έχουν και κάποιο είδους ε, εφαρμογή και θα πρέπει να ταιριάζουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Έχουμε για αγαθά και υπηρεσίες ενιαία αγορά που έχουμε τώρα και για το ανθρώπινο κεφάλαιο, του ανθρώπινου πόρου, μια ενιαία αγορά. Εσά ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τη διαδικασία του Κατσιστιάη, όμω μπορούμε να δώσουμε το λόγο μόνο ει τέσσερι συναδέλφου. Και συγγνώμη, όμω έχω μείνει πάρα πολύ πίσω όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο. Ο, ε, κύριο Μοντέρο, η κυρία Μοντέρο Αγγελιά, συγγνώμη, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Επιτροπέ. Δύο πυλώνες θα πρέπει να στηρίξουν αυτό το θεματολόγιο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε, στα προβλήματα προξενεί το τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές όπου είναι πολύ υψηλή. Και δεύτερον θα πρέπει να ενισχύσει ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές χώρες ε, ως προς την αντιμετώπιση των κενών σε επαγγελματικέ δεξιότητες σε τομείς όπως φερειπίνο τουρισμός που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη και για πολλές χώρες έχει μεγάλο ποσοστό επί του έπτους. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστούν στοιχεία κατάρτισης και αναπόκτησης νέων και κυρίως ψηφιακών δεξιοτήτων για όσο δυνατόν περισσότερους εργαζομένους. Στον τουρισμό πρέπει να δημιουργηθεί ε, να δημιουργηθούν συνθήκες για την ε, κινητικότητα με συνεργασία μέσω μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με μια πλατφόρμα η οποία θα εξασφαλίζει την ε, στήχηση θέσεων εργασίας με δεξιότητες των εργαζομένων και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το έχει πει και το έχει ζητήσει να υπάρχει κοινωνική στρατηγική το Κοινοβούλιο για αυτές τις νέες δεξιότητες. Οπότε είναι θετικό αυτό το θεματολόγιο. Αν δεν θέλουμε όμως να έχουμε νέους φραγμούς και περαιτέρω περιθωριοποίηση για την ψηφιακή κοινωνία. Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τις νέες ευκαιρίες και θα πρέπει να δώσουμε επιγόντως μια νέα όθεση σε αυτού του είδους το θεματολόγιο τους ώστε να αρθούν τα σημερινά κενά και η διαφορά, το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για την ψηφιακή οικονομία. Άρα θα πρέπει να τεθεί επιτάπητο στο πώς θα έχουμε κάποιο είδους αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού του ψηφιακού του, του ίντερνετ να να προχωρήσει να το μάθει ο κόσμος και άρα θέλουμε περισσότερους πόρους για την καταρτήση του ώστε να υπάρχουν εγγύσει ότι οι εργαζόμενοι και ιδίω αυτοί που έχουν λιγότερα προσόντα να αποκτήσουν αυτά που χρειάζεται μια που το περιβάλλον το εργασιακό συνεχώς αλλάζει Κύριε ε, Τόμασης, κύριε Τόμασης, ένα λεπτό. έχουμε τα κράτη τα οποία εντάχθηκαν τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ένα ε, ποσοστό επί του ε, παγκοσμίου ΕΠ πολύ χαμηλό. Πρέπει να γίνουν λοιπόν προσπάθειες για καλύτερη κατάρτιση, για καλύτερες θέσεις εργασίας, για καλύτερη διασύνδεση των δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας. Για να μείνουμε ανταγωνιστικοί πρέπει να προσαρμόσουμε τις ε, δυνατότητες στις νέες ανάγκες. Οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις από τη Netflix και άλλες αντίστοιχες δεν θα μας ε, βοηθήσουν να ε, προχωρήσουμε ο αριθμός των θέσεων εργασίας ε, στην Ευρώπη πρέπει να ενισχυθεί. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Thank Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ελέγξει κάθε τμήμα της ζωής των πολιτών. Θέλετε πρότυπα για δεξιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παιδεία. Τι σημαίνει αυτό απαιτούνται οι ίδιες προϋποθέσεις και προδιαγραφές σε κάθε χώρα. Η ίδια μορφή εκπαίδευσης. θέτα να ελέγξετε τις δεξιότητες που μαθαίνει ο κόσμος και πώς χρησιμοποιούνται αυτές. Όλα αυτά στο κόστος δεκάδων δισεκατομμύριων ευρώ χρημάτων φορολογουμένων. Η παιδεία και η κατάρτιση. Περισσότερα ήταν καλύτερα με λιγότερο κράτος ή λιγότερο υπερκράτος. Λιγότερους πολιτικούς, περισσότερους διδασκάλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ελέγχει τα πάντα, κάθε πτυχή της ζωής. Δυστυχώς. Και χωρίς πρόθεση, αυτό είναι αρνητικό και καταστρεπτικό σε κάθε επίπεδο. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα εν ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Τάισον έχει το λόγο. Έχει το λόγο. Uh, thank you. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και κύριοι, θα είμαι σύντομη στις καταλεκτικές παρατηρήσεις. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ο χρόνος έχει περάσει και η ώρα έχει περάσει και ήμουν άλλωστε και αρκετά διεξοδική στι αρχικέ μου παρατηρήσει. Πάντω, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για τη συμφωνία που καταγράφουμε ω προ την αναγκαιότητα και τη σημασία αυτής της, αυτού των δεξιοτήτων. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με τις μακροοικονομικές ε, πολιτικές ώστε να ενθαρρυνθεί και η δημιουργία θέσεων εργασίας και τα δύο αυτά προχωρούν παράλληλα επί παραδείγματι χάρη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που μας επιτρέπει να δώσουμε με τις επενδύσεις ε, νέα όθηση στις ε, θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις και δει στις θέσεις εργασίας. Η απασχολησιμότητα δεν είναι βρισιά, όπως έχω πει και πιο παλιά. Η κατάρτιση, η εκπαίδευση πρέπει να εκπαιδεύει, να προετοιμάζει τον νέο ώστε να ε, μπαίνει στην κοινωνία ως χρήσιμος πολίτης και πρέπει να του προσφέρει και εγκάρσεις δεξιότητες. Ταυτόχρονα όμως, πολύ σωστά αναμένει ο πολίτης η εκπαίδευση και η κατάρτιση να του, ότι θα του προσφέρει και την ευκαιρία να βρει μια θέση εργασία. Γι' αυτό λοιπόν είναι προς το συμφέρον και της ε, ε οικονομίας αλλά και της προσωπικής ανέλεξης του κάθε ανθρώπου η εκπαίδευση και η κατάρτιση που πρέπει να είναι για όλους για να προστευτούν από την ανεργία και απευθύνεται και σε όλους, ε, ακόμη σε όλους ε, είτε εργάζονται είτε δεν εργάζονται είτε έχουν ιδιαίτερες ε, συνθήκες απασχόλησης είτε έχουν αναπηρίες. Απευθύνεται επίσης το θεματολόγιο σε κάθε έναν εμπλεκόμενο φορέα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα αισθητούτα επαγγελματικής κατάρτισης, τις επιχειρήσεις. Εδώ ανοίγει μια συζήτηση και σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και στα κράτη-μέλη για την υλοποίηση του θεματολογίου. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ για την υποστήριξη, σα ευχαριστώ για την έμπνευση που μα προσφέρετε. Προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σα και όπω είπα και στην εισαγωγική μου παρέμβαση, τα έγγραφα θα είναι στη θέση σα το ταχύτερο δυνατό. Όταν δηλαδή επισήμως εγκριθούν, δηλαδή την προσοχή Παρασκευή, σα ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε Λεώ ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Εδώ πέρα τούτη η συζήτηση. Διότι να ή διακόπτουμε για να περιμένουμε να έλθει ο Υπουργός εκπρόσωπος της υπάτησης εκπροσώπου ή προχωρούμε χωρίς τον εκπρόσωπο της υπάτησης ε, εκπροσώπου.